Ο Πρόεδρος έλαβε την ε, θέση του Συμβουλίου για την πρώτη ανάγνωση σε σχέση με τις ψυχοενεργές ουσίες και τη συμπερίληψή τους στον ορισμό των ε, ναρκωτικών ουσιών. Ο τίτλος αυτός θα ενσωματωθεί στα πρακτικά. Τρεις είναι οι μήνες προθεσμίας που έχει στη θέση του το Κοινοβούλιο και ξεκινά η προθεσμία από αύριο, 6 Οκτωβρίου. 6 Οκτωβρίου 2017. Το κατάλογο λοιπόν θα τον δείτε στα κείμενα.